Βάσει του άρθρου 119 έχω λάβει μια πρόταση μορφής έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1 δέκατο των βουλευτών. Η συζήτηση για την πρόταση μορφής θα γίνει στην επόμενη ε, σύνοδο του Κοινοβουλίου. Έρχομαι τώρα